Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι εργασίες της Ολομέλειας. Παρακαλώ οι συζητήσεις να μην διεξάγονται εντός της Ολομέλειας. Θα ήθελα οι συζητήσεις παρακαλώ στα αγγλικά το λέει η Πρόεδρος να γίνουν εκτός αιθούσης. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη από πλευράς της Αντιπροέδρου της Επιτροπής θα λάβει τον λόγο ο εκπρόσωπος. Παρακαλώ έχετε τον λόγο